χρησιμοποιούσαν αυτά τα υφιστάμενα δίκτυα για να διασυνδεθούν οι γυναίκες στις διάφορες αγροτικές περιοχές. Ε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Έχει σειρά η έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών σταθμών στα νέα κράτη-μέλη. Για τέσσερα λεπτά ο εισηγητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, οι συνθήκες προσχώρησης της Λοβακίας, της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας συμπεριλαμβάνουν τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών που δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας και δεν μπορούν να εξυγχρονιστούν. Στόχος της Ένωσης δεν ήταν να καλύψει συνολικά το κόστος παροπλισμού, αλλά αφορούσε και στην διαχείριση των αποβλήτων, την απορρίπανση των χώρων των εργασιών παροπλισμού και επανόρθωσης και αποκατάστασης συγγνώμη. Βελτίωση επίσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και παρέμβαση στην όλη διαμόρφωση της ενεργειακής ασφάλειας. Επίσης, κατάρτιση του προσωπικού, ασφάλεια του προσωπικού που θα συμμετέχει στη διαδικασία του παρεπλισμού. Αυτά ορίστηκαν χωρίς να έχουμε μία όροφη. Και επειδή δεν είχαμε την οροφή, δόθηκαν επιπλέον χρηματοδοτήσεις της τάξης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σταδιακά εδόθησαν. Το ελεγκτικό συνέδριο ζητά να ξεκαθαριστούν ορισμένες πλευρές του θέματος. Αυτά τα χρήματα δαπανήθηκαν για τον παροπλισμό Υπάρχει ασφάλεια στην εναπόθεση των αποβλήτων. Χρησιμοποιείται η κεκτημένη εμπειρία επαρκώς. Και τα λαμβάνονται υπόψη περασμένα σχέδια για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος. Χρειάζεται περαιτέρω χρηματοδότηση και αν χρειαστεί να δοθεί περαιτέρω χρηματοδότηση για τα ενεργειακά σχέδια θα φτάσει ή πρέπει να επικεντρωθούμε στα σχέδια παροπλισμού. Πιστεύετε όμως ότι αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να συνεχίζονται, να χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο κύριος Νικολάσικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά τον παραπλισμό των ε, πυρηνικών σταθμών στις ε, τρεις χώρες, ε, η χρήση των κρατικών κονδυλίων δεν ήταν επαρκής. Ε, γι' αυτός ε, δόθηκαν ενισχύσεις από την ε, κοινότητα. Οι μελέτες δείχνουν βέβαια ότι το κόστος για τον παροπλισμό το κλείσιμο σήμερα έχουν ξεπεράσει τις ενισχύσεις που είχαν σχεδιαστεί και τις εκτιμήσεις παρόλο που ο παροπλισμός βρίσκεται ακόμα στην πρώτη φάση. Θα πρέπει να συνεχίσει ο παροπλισμός μέσα στα πλαίσια των οικονομικών προοπτικών του 2013. Γι' αυτό θα πρέπει τα μέσα για τον παροπλισμό των τριών ε, πυρηνικών σταθμών να ε, εξευρεθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 143 πυρηνικά εργοστάσια και το Μάρτιο για το 2010 η πυρηνική ενέργεια αποτελεί το 28% του ευρωπαϊκού μίξ. Και αυτά τα λένε οι στατιστικές. Τα γεγονότα στη Ιαπωνία σήμαναν το συναγερμό για το ρίσκο. Το κλείσιμο και ο παροπλισμός των πυρηνικών εργοστασίων αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό βάρος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να χορηγήσει τα σχετικά χρήματα για τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, διότι η έλλειψη κονδυλίων μπορεί να καθυστερήσει τα σχέδια παροπλισμού και αυτό ενηχεύει κινδύνους. Θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν τα σχέδια παροπλισμού και η Κομισιόν επεξεργαστεί και μία έκθεση σχετικά προβλέποντας μία μακροπρόθεσμη χρηματική ενίσχυση για τα σχέδια. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Κύριε Ευχαριστώ. Ε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον συνάδελφο και να ευχαριστήσω για καλή συνεργασία. Έχουν τρεις χώρες μέλη περίπλοκες υποχρεώσεις για το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών. Έχουμε τα οικονομικά μέσα και την ε, αλληλεγγύη υποχρέωση παροχής οικονομικής βοήθειας για το κλείσιμο και για να μετριάσουμε τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν ακόμα, που δεν έχουν διευθετηθεί. Υπάρχει δομή περίπλοκη σε πολλά κράτη-μέλη, ούτως ώστε δεν μπορεί να γίνει απορρόφηση κονδυλίων ε, ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να έχει καλύτερο συντονιστικό ρόλο και να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα κράτη-μέλη έχουν πυρηνικούς σταθμούς ε, στο έδαφος τους. Πολλά από αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια είναι παροχημένα. Ε, πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ώστε θα παροπληστούν κάποια από αυτά για λόγους ασφαλείας και για να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Τα νέα κράτη-μέλη έπρεπε να κλείσουν ε, γρήγορα τα δικά τους ε, πυρηνικά εργοστάσια και έπρεπε να λάβουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει με ασφάλεια αυτός ο παροπλισμός. Αυτό φυσικά ε, δεν πρέπει να θέτει σε κινδύνο την σωστή ε, διάθεση των αποβλήτων, τη σωστή προσαρμογή των εργοστασίων αυτών, των σταθμών αυτών και την ε, σωστή αντικατάσταση της πυρηνικής ενέργειας μάλιστα πηγές ενέργειας. Αυτή η μελέτη λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις κοινωνικές επιπτώσεις όλων αυτών, πέρα από τα θέματα της ασφαλείας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά του παροπλισμού. Ε, δεν είναι μόνο η ασφάλεια των εργαζόμενων, είναι και η δουλειά τους που διακυβεύεται. Για ένα λεπτό κύριο Πάσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου, η οποία έχει να κάνει με τον παροπλισμό ε, των ε, πυρηνικών σταθμών. Στην ε, Σλοβακία μετά το Τσερνομπίλ μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε εξυγχρονισμένη τεχνολογία από τους Γερμανούς και τους Γάλλους. Η Διεθνής Ένωση για την Πυρηνική Ενέργεια διασφάλισε ότι ακόμα για 13 χρόνια θα μπορέσει στη Σλοβακία να λειτουργήσει ο πυρηνικό μα σταθμό. Ε, ε, για να καθισχάσουμε λοιπόν τους αυστριακούς γειτόνους μας ε, θα πούμε ότι βρισκόμαστε στην Πόνιτσα σε μια πολύ καλή φάση. Αυτό σημαίνει ότι ε, προσπαθούμε τουλάχιστον εν μέρη να αντικαταστήσουμε τις απώλειες ε, στη ε, δημιουργία της, την δημοκρατία της Σλοβακίας σε ενέργεια και ανθρώπινες εργασίες. Η Επίτροπος Ρέντινγκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει την εισήγηση για την χρηματοδότηση για την διάλυση πυρηνικών σταθμών. Ξέρετε ότι η πυρηνική ασφάλεια είναι και θα παραμείνει απόλυτη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις προσπάθειες διάλυσης και παροπλισμού για πυρηνικούς σταθμούς που δεν αναβαθμίστηκαν με τρόπο ικανοποιητικό μοιραζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές από τις απόψεις της εισήχησης. Συμφωνούμε για την ανάγκη τα κράτη να υποβάλουν λεπτομερή σχέδια παροπλισμού όπως και έναν προγραμματισμό μακροπρόθεσμο, οικονομικό, χρηματοδοτικό τα κονδύλια θα πρέπει να δίδονται για τις δραστηριότητες διάλυσης και η Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο να παίξει ούτω ώστε να υπάρξει ε, αυστηρή παρακολούθηση των εργασιών. Πιστεύουμε στην υποχρέωση να τηρηθεί η αρχή του ρηπαίνοντος που πρέπει να πληρώνει. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί που χρησιμοποιούν τον πυρηνικό σταθμό, που τον διαχειρίζονται, να εξασφαλίσουν ε, τα κονδύλια κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής του πυρηνικού σταθμού. Θα πρέπει ο πυρηνικός σταθμός να είναι στο δυνατόν πιο ασφαλής και να υπάρχει μια, μια διαφάνεια στις εργασίες παροπλισμού. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το, η εισήγηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον παροπλισμό. Η Επιτροπή θα ήθελε σε διάφορα μέρη της εισήγησης να υπάρξει μια αναγνώριση ότι ο βασικός στόχος της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρώτα απ' όλα να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των μονάδων και να παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί αυτοί για λόγους ασφαλείας. Νομίζουμε ότι ο στόχος αυτός είναι βασικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν, ε, όταν αξιολογείται η αποδοτικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης ποτέ δεν καλύπτει το πλήρες κόστος ε, της, του παροπλισμού, ούτε αντισταθμίζει όλες τις συνέπειες. Η υποστήριξη απλώς συμβάλλει ε, στην αντιστάθμιση της προ, του πρόωρου κλεισίματος. Το κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει την πλήρη ευθύνη για τον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων και είναι ευθύνη του κράτους μέλους να υποβάλει λεπτομερή προγραμματισμό και το κράτος μέλος επίσης πρέπει να υποβάλει χρονοδιάγραμμα λεπτομερές και το κόστος για τον πλήρη παροπλισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την, το Κοινοβούλιο για αυτό την επίκαιρη εισήγηση ε, για το θέμα που με την Φουκουσίμα έχει γίνει ακόμα πιο επίκαιρο. Ε, είναι σημαντική η πυρηνική ασφάλεια. Θέλουμε να έχουμε στο το δυνατόν τους ε, καλύτερους κανόνες και πρότυπα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 Αρίφ για την